Βλέπετε λοιπόν ε, το θέμα αυτό που ε, θα ε, διατυπωθεί στα πρακτικά. Και ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση Ντεχάνε και Κάλφιν